αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι την εθέτηση των πρακτικών, αυτός ο διορισμός θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται. Αφορά την Κοινοβουλευτική Συνέλευση τη Εκπροσώπηση και Ευρωπαϊκή Ένωσης, ο κύριος Ρεντζέλ θα την καταστήσει τον κύριο Ρουάς. La prima...